Επόμενο θέμα στην ημερήσια δέταξη είναι η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο. Όσοι ήθιστε, θα παρακαλέσω τους συναδέλφους που θέλουν να συμμετέχουν στην ώρα των ερωτήσεων να έρθουν προς τα εμπρός αν θέλουν, να κατεβούν στα την έδρανα. Και η πρώτη ερώτηση είναι του κυρίου Πόσελτ και αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα. Κυρία Μάλσον, όποτε θέλετε έχετε το λόγο. I am of ready to move. Ευχαριστώ, βεβαίω. Να πάω από τι Ηνωμένε Πολιτείε στην Κούβα. Δεν είναι ένα πρόβλημα. Κύριε Πόσελ, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, ανησυχεί βαθύτατα το Συμβούλιο πάντοτε για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, ιδιαίτερα ε, την έλλειψη πρόοδου για πολιτικά και ε, ατομικά δικαιώματα. Οι Κουβανοί δεν έχουν ελεύθερη έκφραση, ελεύθερο τύπο και δικαίωμα στο συνέρχεστε. Περιορισμός και στο ίντερνετ, περιορισμός της ελευθερίας των πολιτών, στην είσοδο του στη χώρα και στην ε, κυκλοφορία τους. 8 ε, είναι οι πολιτικοί κρατούμενοι, 34 το 2000 ήταν, αλλά ε, είναι προς το τέλος της ποινής τους παρατηρείται η κατάσταση και υπάρχουν και αντίστοιχες ομάδες παρακολούθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κατάσταση στις φυλακές, σύμφωνα με ε, δηλώσεις των πολιτικών κρατουμένων οικογενειών και άλλων οργανώσεων, είναι πολύ κατώτερες και υπολοιπόμενες ε, των διεθνών ε, προτύπων πολλοί δεν έχουν και την ιατρική περίθαλψη που πρέπει να έχουν όπως λένε οι τους. Ε, είναι ε, ταπεινωτική η συμπεριφορά προς αυτούς, ε, ψυχολογική πίεση μέχρι και σωματική βία. Ωστόσο δεν έχουν διωχθεί ούτε φυλακές ούτε αστυνομικοί. Η Κούβα αρνείται ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι και δεν δέχεται έλεγχο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από ανεξάρτητες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο έχει στην προσέγγιση του μια κοινή θέση ε, του 1996 για την Κούβα και Έκτοτε ετησίως ε, αξιολογείται αυτή η θέση. Τον Οκτώβριο του 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κούβα συμφώνησαν να αρχίσουν ένα ευρύτατο και εκτενέστατο πολιτικό διάλογο σε σχέση και συνάφεια με τις κοινοτικές πολιτικές και όχι μόνο με τις αρχές της αλλά και με τη δημοκρατική αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών. Ε, μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα των ελευθεριών ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στην ετήσια αξιολόγηση της κοινής θέσης του 2009. Ολοκληρώνοντας τα συμπεράσματα φέτος τον Ιούνιο, ξεκαθαρίσαμε ότι τα θέματα θα παραμείνουν βασικές προτεραιότητες στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Κούβας. Καλούμε ιδιαιτέρως να απελευθερώσει η κουβανική κυβέρνηση όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που συνελήφθησαν το 2003 και εκφράζουμε ανησυχίες για την κατάσταση της υγείας των πολιτικών κρατουμένων. Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί τις αρχές της Κούβας να ε, αφήσουν αμέσως ε, να μπουν στις φυλακές εκπρόσωποι οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από το προηγούμενο περσινό διάλογο η ευρωπαϊκή πλευρά σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε συνεδρία συμφέρει το θέμα των πολιτικών κρατουμένων. Και σύμφωνα με τα τελευταία συμπεράσματα του Συμβουλίου θα πρέπει πάντα σε επισκέψεις τέτοιου υψηλού επίπεδου να ασχολούμαστε με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να συναντούμε ειρηνικού ε, δημοκρατικούς εκπροσώπους της αντιπολίτευσης. Είναι σημαντικό να έχουμε διάλογο με την Κούβα γιατί έτσι ειλικρινά μπορούμε να συζητούμε θέματα ε, αμοιβαίου ενδιαφέροντος και ανησυχίας. Μεταξύ αυτών και η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο ανησυχούμε βαθύτατα ακόμα και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με μονομένες περιπτώσεις ιδιαίτερα κρατουμένους με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα ε, την κατάσταση ενός κρατουμένου που αναφέρεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε την αλληλεγγύη της ε, την Σουηδική Προεδρία στην Αβάνα τον Αύγουστο. Έγινε μια διαδήλωση για να δείξουμε στην οικογένεια του ιατρού κυρίου ε, Ντάρση Φερέρα ότι ανησυχούμε και ότι παραβιάζονται τα δικαιώματα του από τις κουβανικές αρχές. Και ο κύριος Αλφρέντο Δομίνγκες, ο άλλος κρατούμενος, επίσης είναι κάτι που μας απασχολεί και ε, το θέτουμε υπόψη των κουβανών στους διαλόγους που έχουμε και είμαστε και σε επαφή με την οικογένειά του. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρα. Ευχαριστώ κύριο Σπόσελτ. Ναι, θα ήθελα να πω στην Προεδρεύουσα ότι την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η απάντησή τη, πάρα πολύ εμπεριστατωμένη. Η διεθνή Κοινότητα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με έχει ενημερώσει για το πώ έχουν οι συνθήκε κράτηση στην Κούβα και θέλω να ρωτήσω πρώτον, το Συμβούλιο πραγματικά μπορεί να ε, ε, ελέγξει πώ κρατούνται και πώ ζουν οι διάφοροι κρατούμενοι και μετά πώ αξιολογεί τι εξελίξει στην Κούβα το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τι σχέσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση.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 αξιότιμοι βουλευτά, δεν έχουμε πρόσβαση επίσημα σε τέτοιες πληροφορίες, αλλά μέσω διεθνών οργανισμών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, επαφών, πολιτικών ε, ομάδων, ε, παίρνουμε κάποιες τέτοιες ε, κατακαιρματισμένες όμως πληροφορίες για την κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων και ξέρουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σοβαρά τα προβλήματα υγείας που έχουν. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τις οικογένειες και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις για να διευκολύνουμε την κατάσταση, αλλά τι να κάνουμε δεν έχουμε. Έχουμε λιγοστές ε, και αναξακρύβωτες πληροφορίες. Πολλοί από αυτούς τους κρατούμενους ε, δεν έχουν δικαστεί, δεν, ε, δεν τους έχει καν απαγγελθεί η κατηγορία. Δηλαδή αυτό αντιβαίνει ακόμη και στην νομοθεσία της Κούβας. Δικαιούνται να μάθουν γιατί είναι στο, στη φυλακή και βασικά τι, γιατί πράγμα να τους κατηγορούν. Αλλά τι να κάνουμε που έχει έτσι η κατάσταση στην Κούβα. Ε, ε, ε, ο διάλογος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερες δυσκολίες αλλά παρόλα αυτά, ε, καλό είναι να διατηρηθεί ε, αυτός ο διάλογος, γιατί χάρη σε αυτόν έχουμε τη δυνατότητα να ερχόμαστε σε κάποια επαφή με τις αρχές και να δείχνουμε, να απευθύνουμε σκληρές επικρίσεις, αλλά να ερχόμαστε και σε επαφή με τους αντιφρονούντες και την ε, κοινωνία των πολιτών, τους ειρηνικούς αντιφρονούντες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Προς το παρόν, τι είναι η ρότα που νομίζουμε πρέπει να ακολουθήσουμε και στο προσεχές μήνα δεν προβλέπεται αλλαγή. Ε, σας ευχαριστούμε. Ε, ε, δύο επερωτήσεις. Θα ακούσουμε τις επερωτήσεις και μετά θα τις απαντήσει ε, η ε, Προεδρεύουσα, ο κύριος Χουντής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. κυρία Υπουργέ, επειδή πιστεύω ότι και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπω αυτά τα θέματα που θέτει ο συνάδελφο Πόσελτ με την ερώτησή του μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα με χώρε με τι οποίε έχουμε πολιτικέ διπλωματικέ σχέσει και οικονομικέ συναλλαγέ μου προκαλεί εντύπωση το γεγονό ότι η ευρωπαϊκή ένωση και τα κράτη μέλη τη κρατάνε παθητική έω αρνητική στάση απέναντι στο λογικό και πάγιο αίτημα τη δημοκρατία τη κούβα να αρθεί ο αποκλεισμό του από τι ηνωμένε πολιτείε. ερωτώ λοιπόν πώ βλέπει το θέμα η προεδρία και πώ νομίζετε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα από τα κράτη μέλη εν ώψη του γεγονότο ότι η κούβα καταθέτει όπω είναι γνωστό στη γενική συνέλευση του οηε στι 28 δεκάτου σχετικό ψήφισμα για να αρθεί ο αποκλεισμό τη από τι ηνωμένε πολιτείε. σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία για την ώρα. Ηνωμένε Πολιτείε. Ναι, ξαναρχίζω. Εδώ είμαι μια ειρηνική αντιφρονούντα από ένα από τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ουγγαρία. Ήθελα τη δική σα συμβουλή. Πώ να επιτύχουμε το ίδιο επίπεδο ενδιαφέροντος για την κατάσταση ανθρωπινών δικαιωμάτων και στην Ουγγαρία, όπω αυτό που δείχνατε για την Κούβα. Διότι στην Ουγγαρία από το φθινόπωρο το 2006 έχουμε αστυνομικές διώξεις και ξυλοδαρμούς κατά διαδηλωτών βασανιστήρια στις φυλακές. Με συγχωρείτε, ξεπέρασα 30 δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, θέλω να ρωτήσω, ε, οι κουβανοί πολιτικοί μπορεί να διαπραγματευτούν εκ μέρους μας. Εκτός μικροφώνου πάλι ομιλήτρια. Με συγχωρείτε, 30 δευτερόλεπτα έχετε και το ερώτησή σας αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κούβα. Υπουργέ, θέλετε να απαντήσετε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλέ ε, ευκαιρίε έχει εκφραστεί κατά του Αμερικανικού εμπάργκο. Νομίζουμε ότι δεν διευκολύνει σε τίποτε την εξέβρεση κάποια λύση για την Κούβα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προ στιγμή έχει εκφράσει την προθυμία τη να έχει στενότερη συνεργασία με την Κούβα, ε, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, αλλά ανάλογα με την πρόοδο που θα επιτελέσουν εκείνοι στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έλλειψη πρόοδου στα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, ο σεβασμό τη δημοκρατία η έλλειψη σεβασμού στη δημοκρατία και ο αριθμό των πολιτικών κρατουμένων δεν μα επιτρέπουν να επιτελέσουμε πρόοδο στον τομέα αυτό. Πρέπει οι κουβανοί να μα δείξουν ότι θέλουν τέτοια σχέση μαζί μα και ότι μπορούν να επιτύχουν χειροπιαστή πρόοδο, χειροπιαστά αποτελέσματα στον τομέα αυτό. Αυτό για την ώρα είναι μάλλον αμφισβητήσιμο. Σα ευχαριστούμε. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Την κυρία Χάρκιν. Αφορά την κακομεταχείριση υπερηλίκων. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να παραμείνετε στο χρόνο που προβλέπουν οι κανόνες για την ερώτησή σας. 30 δευτερόλεπτα. Παραμείνετε στο θέμα της ε, προβλεπόμενης ερώτησης. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση όπου έτοιμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Χαρκέν. Ε, μας έθεσε ένα ερώτημα εξαιρετικά επίκο, επίκαιρο για ένα, γιατί ε, λόγω του γυράσκοντος πληθυσμού ε, και φυσικά είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας ως επιτοπλίστων και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει και να συμπληρώσει μόνο τη δράση των κρατών μέλων. Η Σουηδική Προεδρία θα ήθελε να εστιάσει την προσοχή της σε αυτό το θέμα για να αναβαθμίσει την ποιότητα των υπηρεσιών στον τομέα της υγείας για τους ηλικιωμένους και να καταπολεμήσει την κακοποίηση των ηλικιωμένων ηλικιωμένων. Έγινε και μία διάσκεψη πριν από ένα μήνα στη Στοκχόλμη ε, για την αξιοπρεπή και υγιή γύρανση 160 άτομα από 27 διαφορετικά κράτη. Ε, υψηλό επίπεδο προσέλευσης εκπροσωπήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη, διάφοροι υπάλληλοι Υπουργείων Υγείας ε, και πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Ο Στόχο ήταν ακριβώς να υπάρξει ευαισθητοποίηση για αυτά τα ζητήματα που μιλάει και η κυρία Χάρκιν. Δηλαδή πώς μπορούμε να χειριστούμε ε, αυτό, αυτή την πραγματικότητα. Δηλαδή θα, θα χρειαστεί μια ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της υγείας και τη παροχή παροχής υγειονομικής φροντίδας για να καλύψουμε τις ανάγκες ε, των ηλικιωμένων. Ε, θα, Στι 30 Νοεμβρίου στο, στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα εγκριθούν σχετικά συμπεράσματα και το σχέδιο συμπεράσματων ε, το τονίζει ότι χρειάζεται εγκύτερη εντονότερη συνεργασία στον τομέα ε, τη υγιού και αξιοπρεπού γύρανση, ε, μεταξύ άλλων μέσω τη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και θα είναι την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει σχέδιο δράση για την αξιοπρεπία και την ποιότητα ζωή των ηλικιωμένων. Σα υπενθυμίζω επίση ότι ενέκρινε τον Ιούνιο συμπεράσματα το Συμβούλιο για την ισότητα των ευκαιριών για τους άντρες και τις γυναίκες στην αξιοπρεπιακή γύρανση για να έχουμε υψηλού επίπεδου υπηρεσίες για τη φροντίδα των ηλικιωμένων ε, στα διάφορα ιδρύματα και ε, για την οικιακή φροντίδα. Ε, σχετικά τώρα με την κακοποίηση των ηλικιωμένων πιο συγκεκριμένα, ο κανονισμός του Συμβουλίου υπαριθμών 78 του 2008 απαγορεύει την διακριτική μεταχείριση λόγω ηλικία στο χώρο εργασία και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρυνθεί η προστασία, ώστε να καλύψει και άλλους τομείς, η κοινωνική προστασία, τομέ της υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, πρόσβαση στις υπηρεσίες, στέγαση κτλ. Αυτή η πρόταση καλύπτει πολλά σχετικά τμήματα όπου αναφέρεται το θέμα της κακοποίησης ε, των ηλικιωμένων ε, και στο σπίτι και στα διάφορα ιδρύματα ε, του τομέα της υγειονομικής φροντίδας. Ακόμη και παρενόχληση είναι μια μορφή διακριτικής μεταχείρισης και να παραθέσω εδώ τον ορισμό δηλαδή παραβιάζεται η ακαιρεότητα του ατόμου και υφίσταται με μία ε, ταπεινωτική, επιθετική και αρνητική συμπεριφορά. Και αυτό συζητείται στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη εγκρίνει το ψήφισμά του. Βέβαια, ε, στο Συμβούλιο χρειάζεται ομοφωνία. Ε, δεν μπορώ να προδικάσω το αποτελέσμα των συζητήσεων στο Συμβούλιο. Θα ήθελα να πω ότι καταβάλουμε τι προσπάθειε που μπορούμε, ούτω ώστε νομοθετικώ πω να υπάρξει ρύθμιση για να καταργηθεί οποιαδήποτε αρνητική μεταχείριση και κακοποίηση των ηλικιωμένων βάσει του ψηφίου μα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κανένα άνθρωπο δεν πρέπει να υφίσταται τέτοιε παρενοχλήσει, τέτοιε κακοποίησει και κυρίω όχι ε, οι ηλικιωμένοι μα που εξαρτώνται από εμά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ την κυρία Μάνστρομ για την ιδιαίτερα απάντησή τη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τη Επιτροπή από το 2008, οι καλέ συνθήκε πρέπει να προλευθούν, κατάλληλε συνθήκε πρέπει να προσταθούν για την σπόρου και την κατάρτιση και την ε, λειτουργία των ε, υπευθύνων για του υπερήλικε. Είναι ένα από του τομεί όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει δράση. Έχει διασυνοριακέ διαστάσει. Ήθελα λοιπόν να ξέρω την άποψή σα για τη θέσπιση μια επίσημη δομή για την ανταλλαγή πληροφοριών σε ό,τι αφορά του επαγγελματίε του τομέα υγεία. Ιδίω όσου εργάζονται και διασυνοριακά. Σα ευχαριστούμε κυρία Υπουργέ. Κυρία Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ για αυτή την πρόταση. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, για να είμαι ειλικρινή. Ακούγεται μια πολύ καλή πρωτοβουλία, αλλά θα πρέπει να ναι. το συζητήσω με του υπόλοιπου υπουργού και να το θέσω επιτάπητο. Ίσως θα μπορούσαμε να το ξαναδούμε κάπως αργότερα, αν δεν σας πειράζει. Ευχαριστούμε. Και πάλι δύο συμπληρωματικέ ερωτήσει με τη σειρά. Η κυρία Τσίκαου πρώτη. Uh, κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, οι λαοί ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βλέπουμε ότι ε, αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο κοινωνικό λοιπόν αυτό πλαίσιο, ποιες είναι συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν κάνει τα κατημέλη για να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής των υπερελληνικών. Ευχαριστώ. Okay, Mr. Kelly. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ η κυρία Χάρκιν έκανε μια πολύ σημαντική ερώτηση και πολύ ωραία την απαντήσατε. Διευρύνοντας λίγο το πεδίο. Σήμερα ηλικιωμένοι είναι ότι ε, είναι πάνω από 65 ετών όλοι οι άνθρωποι. Σκέφτεστε να έχουμε μια μετάβαση προς μια πιο προοδευτική συνταξιοδότηση και όχι στα 65 έτσι να διακόπτεται απότομα, αλλά σταδιακά βαθμία να βγαίνει ο κόσμος στη σύνταξη. Ε, αυτό ξεπερνάει λίγο τον τίτλο της ερώτησης, λέει η Πρόεδρος, αλλά το αφήνω στη διακριτική ευκαιρία της Υπουργού, αν θέλει να το απαντήσει. Ευχαριστώ να απαντήσω στο πρώτο, στην πρώτη ερώτηση. Αυτή, αυτά τα ζητήματα πρέπει να συζητηθούν. Το τρίο, η Γαλλική, Τσεχική και Σουδική Προεδρία συμφωνήσαμε να ενισχύσουμε διάλογο για ζητήματα που έχουν σχέση με την υγεία και τι υπερήλικε. Έγινε σύνοδο για το Αλσχάιμερ, αν θυμάστε, και σύνοδο που <coughs> ανέφερα και εγώ το προηγούμενο μήνα για τι εξωπρεπεί συνθήκε διαβίωση και την εξωπρεπή μεταχείριση των υπερήλικων. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία να συζητήσουμε τέτοια θέματα. Τα συμπεράσματα μάλιστα θα παρουσιαστούν στην ΕΠΣΚΟ το τέλο Νοεμβρίου. Και εκεί θα δούμε και την έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά για την ηλικία συνταξιδότηση. Αυτό είναι κάτι που αποφασίζει κάθε κράτο μέλο για τον εαυτό του. Όμω η συνθήκη που είχαμε στα πλαίσια τη στρατηγική τη Λισαβόνα, όχι τη συνθήκη για μια φορά, τη στρατηγική τη Λισαβόνα, για το πώ να έχουμε την οικονομική ανάπτυξη, τι δυνατότητε οικονομική ανάπτυξη, την απασχολησιμότητα, τι γεωγραφικέ προκλήσει σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα. Να ένα σημείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη για να εκμεταλλευτούμε και την αρμοδιότητα και την εμπειρία των υπηρελικών να μείνουν εντό τη εργατική δύναμη. Όμω αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει μόνο το Συμβούλιο. Δεν μπορεί να θέσει μια ηλικία όριο για αυτή τη σύνταξη. Τα επιμέρου κράτη-μέλη εδώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν όπω θέλουν την εργατική του δύναμη. Ευχαριστούμε. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση. Από τον κύριο Σμιτ. Για τον Σουηδό δημοσιογράφο, τον κύριο Ντάιβιτ Άιζακ, που κατέται σε φυλακή, τη Ερυθρέα. Υπουργέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να βρω το σωστό χαρτί. Ένα λεπτάκι. Οχτώ χρόνια έχουν περάσει από τότε που ο Σουηδοερυθρέος ε, δημοσιογράφος Νταβίτ ε, Ισακ ε, μπήκε στη φυλακή της Ερυθρέας χωρίς να το έχει απαγγελθεί κατηγορία, χωρίς να έχει δικαστεί διάφορες και κανείς δεν μπορεί να τον επισκεφθεί ούτε η οικογένειά του ούτε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ερυθρέα δυστυχώς δεν έχει κανένα καλό ιονό για το μέλλον και η κυβέρνηση της Ερυθρέα είναι η μόνη που μπορεί να κάνει κάτι. Δεν είναι τηρή τι υποχρεώσει τη ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βάσει του διεθνού δικαίου, αυτό είναι πηγή μεγάλη ανησυχία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίω ε, για του ε, πολιτικού κρατουμένου και για την κατάργηση τη ελευθερία έκφραση. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, άνεφόρων στην Ερυθρέα και φυσικά και του συγκεκριμένου δημοσιογράφου. Τον περασμένο περασμένο Σεπτεμβρίο έγινε μια σαφής δήλωση όπου επαναλάβαμε να απελευθερωθούν ανεφόρων όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι και διαπιστώσαμε ότι παραβιάζονται σαφώς οι υποχρεώσεις της Ερυθρέας βάσει τη συμφωνία του ΟΗΕ, της σύμβασης του ΟΗΕ, συγγνώμη, για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει επικυρώσει η Ερυθρέα. Ε, θα πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα αυτό το θέμα για την Σουηδική Προεδρία, για τη Σουηδική Κυβέρνηση και για την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες ε, μέχρι να απελευθερωθεί ο δημοσιογράφος για ανθρωπιστικού λόγου, ε, και να επανενωθεί με την οικογένειά του. Και φυσικά πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, όχι μόνο η δική του κατάσταση, αλλά η κατάσταση γενικώ των πολιτικών ε, κρατουμένων. Στα πλαίσια των σχέσεων ΕΕ και Ερυθρέα, ε, θέλουμε να ισχύσουμε τη συνεργασία για να βελτιώσουμε την κατάσταση ω προ τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό είναι συνάρτηση τη Συμφωνία ε, Κοτονού. Και εκεί πέρα αναφέρεται και το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το θέμα του πολιτικού διαλόγου, ώστε να επιφέρουμε κάποια αλλαγή. Αυτή η προϊούσα διαδικασία είναι απελπιστικά αργή, αλλά ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο και τελικά θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Συγγνώμη. Ε, ο κύριο Σμιτ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για την απάντηση. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω περαιτέρω την ε, ε, χείριστη κατάσταση του δημοσιογράφου. Μας την περιέγραψε καλά η κυρία Μάλμστρομ αλλά ήθελα να μάθω. Ε, ε, ε, δηλαδή, άσκησε το δικαίωμά του να εκφραστεί ελεύθερα και κρατείται στην Ερυθρέα. Δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ειδική δήλωση για τον Ντέβιτ Ίσακ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν πρέπει να κάνει ειδική δήλωση και η Υπουργό Μάλμστρομ ή κάποιο άλλο δεν πρέπει να μεταβεί στην Ερυθρέα για να προσπαθήσει να ε, συναντήσει τον κρατούμενο και τον πρόεδρο Αφεβέρκη. Ε, θεωρώ ότι είναι παράλογο ένα πολίτη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή τόσα χρόνια να είναι μέσα στη φυλακή χωρί δίκη και μπορεί να πεθάνει στη φυλακή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Ούλε Σμιτ, ε, ε, φυσικά συμφωνώ με την απογοήτευσή σου και την ανησυχία που εξέφρασε. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνία με την κυβέρνηση τη Ερυθρέα. Ο Όλε Σμιτ και άλλοι συναδέλφοι έχουν δει ντοκιμαντέρα από την Ερυθρέα, έχουν δει ότι δεν είναι απλέ οι σχέσει με τον πρόεδρο τη Ερυθρέα. Είναι σοβαρά τα προβλήματα που υπάρχουν στι σχέσει μα. Χρησιμοποιούμε του διάβλους που γνωρίζουμε, αλλά δεν έχουμε πρόσβαση πρόσβαση στη φυλάκη. Δεν μπορούμε να τον επισκεφτούμε, τον κρατούμενο. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Ε, Προς το παρόν ε, δεν υπάρχει ε, καμία δυνατότητα για να ασκήσουμε κάποια πίεση, για να τον επισκεφτούμε ή τέλος πάντων να γίνει διάλογος για τον Ντάβιτ Ίσακ ή τουλάχιστον να συναντούμε και με την οικογένειά του που είναι επί του τόπου. Είναι πολύ απογοητευτικό για τη δήλωση που είπε όλοι, όλες Σμίτ ε, από όσο ξέρω είναι ο μόνος ε, ε, κρατούμενος στην Ερυθρέα για αυτούς τους λόγους και πρέπει να δώσουμε στην Ερυθρέα να καταλάβει ότι δεν μπορεί να καταπατά την ελευθερία έκφρασης και πρέπει να απελευθερώσει τον δημοσιογράφο βάσει των διεθνών συμβάσεων που έχει επικυρήσει. Προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε έναν κανονικό διάλογο με αυτή τη χώρα. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν επερωτήσεις, ε, οπότε περνάμε στην επόμενη ερώτηση της κυρίας Χέντε σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την κατανάλωση υνοπνεύματος. Υπουργέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Χέντ. Ε, αρχίζοντας, ε, να, σας υπενθ... να υπενθυμίσω στην κυρία Χέντ ότι η Σουηδική Προεδρία ε, έχει θέσει αυτό το θέμα ως βασικό στόχο για την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, στηρίζει τα κράτη-μέλη για να μειωθούν οι ζημιές που σχετίζονται με την κατανάλωση του υνοπνεύματος. Είναι ε, ύψιστη προτεραιότητα για την Προεδρία και έγιναν τρία, ε, τρεις βασικές κινήσεις. Ε, άτυπη συνάντηση τον Ιούλιο στο Γιον των Υπουργών Υγείας ε, όπου τονίστηκε η ε, θέση σε εμπορία των πνευματούχων ποτών και πώς αυτό επηρεάζει την κατανάλωση του ινοπνεύματος ε, κυρίως τους νέους. Επίσης, διάσκεψη προγνωμόνων ε, στις 21 και 22 Νοεμβρίου στη Στοχόλμη, ούτως ώστε να έχουμε βιώσιμη μακροπρόθεσμη και σφαιρική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το ινόπνευμα. Περίπου 450 άτομα από πολλές χώρες συμμετείχαν στη διάσκεψη και υπήρξε υποστήριξη των στόχων της προ ε, ε, Τρίτον, ε, ε, παγκόσμια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου για τον τομέα της υγείας συνδιοργανώθηκε με τη Σουηδική Προεδρία και το ΣΥΝΤΑ που είναι η Επιτροπή για την Αναπτυξιακή Βοήθεια και το Υπουργείο Υγείας της Νορβηγίας και χρηματοδοτήθηκε από διάφορες διεθνείς οργανώσεις ε, συζητήθηκε το θέμα της παγκόσμιας ε, στρατηγικής ε, που θα αρχίσει να ισχύει το Μάιο του 2010 και παρουσιάστηκαν νέες ιδέες για την αντιμετώπιση των ζημιών που σχετίζονται με κατανάλωση του υνοπνεύματος και άλλα θέματα όπως, για νόσους, παραδείγματος χάρη όπως το AIDS, η φυματίωση, ε, και ε, ρωτάτε εδώ αν η Σουηδική Προεδρία θα κάνει κάτι για να γίνει σύντομα αξιολόγηση. Ναι, μα θεωρούμε ότι ήδη έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα και αναγνώρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 ότι ε, το ενόπνευμα είναι βασική απειλή για την δημόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα έχει ευθύνη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει την υπερβολική κατανάλωση του Ε, και αυτό αναφέρθηκε και στα συμπεράσματα των των Υπουργών Υγεία του Νοεμβρίου του 2006. Ε, το 2007 παρακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την κατανάλωση του νοπνεύματο και τι ζημίε που προκαλεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έχουν ε, ε, αλλά δεν έχει περάσει αρκετός καιρός για να αξιολογήσουμε ολόκληρα τα αποτελέσματα στον τομέα της υγείας που έχει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη διάσκεψη των εμπειρογνωμόνων πριν από δύο εβδομάδες έγινε μια ενδιάμεση έκθεση παρουσιάστηκε η ενδιάμεση έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση. Περιμένουμε την τελική έκθεση η οποία όμως αναμένεται για το 2012. Φυσικά η Σουηδική Προεδρία θα εξετάσει τα πορίσματα συμπεράσματα της διάσκεψης των εμπειρογνωμών για το αλκοόλ και τη δημόσια υγεία. Επίσης χρηματοδοτήσαμε διάφορες νέες έρευνες, μελέτες ε, και ε, γνωρίζετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα αυτό το ζήτημα που προανέφερα, δηλαδή πώς η θέση σε εμπορία του υνοπνεύματος και των υνοπνευματούχων ε, ποτών επηρεάζει την κατανάλωση του υνοπνεύματος για τους νέους και για τους ηλικιωμένους και επίσης συντήθηκε και το θέμα των εθνικών πολιτικών στον τομέα αυτό. Ε, για ε, υπάρχει το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου που τώρα ζητείται στην ομάδα εργασίας ε, του Συμβουλίου και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη φάση των εργασιών μας ε, γιατί χρειάζεται να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική και μετά το 2010 όταν θα εκπνεύσει η τωρινή πολιτική και η Σουηδική Προεδρία να μην εγκριθούν ε, το Δεκέμβριο του 2009 τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ε, κοινοτική πολιτική στον τομέα αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Χέι. Ευχαριστώ. Ε, Υπουργέ, ξέρω ότι η Σουηδική Προεδρία έχει διοργανώσει πολύ ωραίες διασκέψεις και ότι είχε αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το ζήτημα. Απλά, ε, εγώ ρώτησα ε, κάτι για την στρατηγική και το ίδιο ρώτησα και πριν από έξι μήνες και μου απαντήσατε ότι πριν το καλοκαίρι θα γινόταν αξιολόγηση της πολιτικής και γι' αυτό ε, υποβάλλω και πάλι την ερώτηση γιατί δεν έχει γίνει η αξιολόγηση. Έχουν συμβεί πάρα πολλά από το 2001 που πρότεινε η τότε Σουηδική Προεδρία τη στρατηγική, εγκρίθηκε η στρατηγική το 2006 και πολλά έχουν γίνει στο μεταξύ. Έχουν αυξηθεί τα ηλικιακά ωραία σε πολλά κράτη-μέλη, έχουν επιβληθεί φόροι για την κατανάλωση υνοπνεύματος κτλ. κτλ. Χαίρομαι χαίρομαι ιδιαίτερα Απλά ήλπιζα ότι θα είχε κάνει ε, ένα μεγαλύτερο βήμα η Σουηδική Προεδρία, αλλά χαίρομαι που έγινε αυτή η διαφήμιση τουλάχιστον για την ε, κατανάλωση του ινοπνεύματος κυρίως ε, στους νέους. Σας ευχαριστώ. Ναι, προσπαθούμε να δώσουμε, να προβάλλουμε το θέμα και να βελτιώσουμε το χρονοδιάγραμμα για να συντονίσουμε τις διάφορες δράσεις που υπάρχουν και για τις δράσεις επερχόμενης Προεδρίας. Ε, ε, σας μίλησα για την ενδιάμεση έκθεση. Ε, έχει σημασία και εμείς και αναλύουμε ε, τη, τα, την, τα αποτελέσματα, τα πορίσματα της διάσκεψης των εμπρογνωμών, Τελικά η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί το 2012. Αλλά τουλάχιστον αυτό που έχουμε καταφέρει είναι ότι έχουν ευαισθητοποιηθεί όλοι σε όλα τα κράτη-μέλη για τα προβλήματα της κατανάλωσης του αλκοόλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Έχουμε δύο ερωτήσεις. Θα ακούσουμε μια με την άλλη. Κύριε Παλέκης, πρώτος. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, πολλοί είναι αυτοί που πέφτουν θύματα τροχαίων ατυχημάτων στους δρόμους του τηλεφόρου της Ευρώπης. Και πολλές φορές αυτό οφείλεται στην κατανάλωση νοπλαπατοδών. Σε πολλές όμως χώρες έχουμε και ψηλό ποσοστό αυτοκτονιών, όπου πάλι ευθύνεται το ενόπνευμα και κατανάλωση ενόπνευματοδών. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν να λάβει αυστηρότερα μέτρα κατά τη κατανάλωση ενόπνευματο ενόπνευματοδών, ιδίω να έχουμε υπόψη τι σκανδιναβικέ πρωτοβουλίε. Ε, μια απαγόρευση λόγω χάρη τη πώληση ε, αλκοόλ σε νέου ανθρώπου. Thank you, eh, Madam President, and thank you, um, eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, Υπουργέ. Ευχαριστώ την κυρία Χέτ που έθεσε το θέμα αυτό στη σκοτία και θέλω να επιστρέψω την προσοχή στο Υπουργό στο θέμα αυτό, ε, γίνεται συζήτηση στην Κοινοβουλία για την ελάχιστη τιμή των ενοπνευματοδών. Ήθελα λοιπόν να δράξω την ευκαιρία για να ζητήσω, να ζητήσω την Υπουργό να μου πει εάν υπάρχει καμιά σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο για μια ελάχιστη τιμή για τα υνοπνευματόδη προϊόντα. Είναι μια τεράστια συζήτηση αυτή τη στιγμή αυτή τη σχολεία. Ήθελα λοιπόν την άποψη του Συμβουλίου, αν του έχει περάσει καν από το μυαλό μια τέτοια ιδέα. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας αυτές. Μία από τις πέντε ενότητες και προτεραιότητες ακριβώς είναι η μείωση ε, των τραυματιών και των θανάτων ε, στα τροχέα ε, που οφείλονται στο ενόπνευμα και προκαλούν τεράστια οδύνη και οικονομικό κόστος. Συστήσαμε λοιπόν ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα ελάχιστο όριο για νέους ε, άπειρους ε, ερασιτέχνες οδηγούς. Υπάρχει μια σύσταση τέτοια λοιπόν και συνεργαζόμαστε και με τα κράτη-μέλη που ήδη εφαρμόζουν αυτή τη σύσταση και γενικά αυξάνεται η συνειδητοποίηση του κοινού για το θέμα αυτό. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα για τις συζητήσεις που γίνονται σχετικά με την τιμολόγηση Μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο, θα το συγκρίνω και θα το ρωτήσω τον Υπουργό Υγείας που είναι αρμόδιος. Αυτό το συγκεκριμένο θέμα δεν το έχουμε συζητήσει για τις τιμές της ελάχιστες, προς το παρόν τουλάχιστον, διότι δεν είναι και κοινοτική αρμοδιότητα άλλωστε. Ευχαριστώ η Πρόεδρος και τώρα προχωρούμε στην επόμενη ερώτηση του κυρίου Παλέκης με θέμα περιβαλλοντική διάσταση των αγωγών φυσικού αερίου. Παρακαλώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ. North Stream. Είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα για τη Βαλτική θάλασσα λόγω μεγέθους και λόγω πιθανόμενων επιπτώσεων. Ε, το ε, Συμβούλιο γνωρίζει όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και το Nord Stream και λαμβάνει υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις επιπτώσεις ε, προς το περιβάλλον για τη συμφωνία με τη Ρωσία που εγκρίθηκε τον περασμένο Ιούλιο. Όλα τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλη στη σύμβαση του ΕΣΠΟ ε, του 1991 σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων για το περιβάλλον σε διασυνοριακό πλαίσιο ε, και υπάρχουν ε, δεσμευτικές υποχρεώσεις ε, για τους εταίρους ούτως ώστε να γίνεται αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενός προγράμματος. Στη Βαλτική θάλασσα το προσχέδιο Nord πρέπει να εξεταστεί με πάσα σοβαρότητα και πρέπει να δούμε το θέμα επίσης των χημικών ε, και των ορυχείων τώρα. Η χλωρίδα και η πανίδα μπορούν να επηρεαστούν σοβαρά και ο αγωγός φυσικού αερίου βρίσκεται σε σημαντικούς θαλασσίους διάβλους και αυτό συνεπάγεται κινδύνους. Ε, όλες ε, οι χώρες της Βαλτικής εδώ και τρία χρόνια συνεργάζονται ε, για να επομιστεί ο καθένας τις ευθύνες του σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος Nord Stream. Είναι υπεύθυνη μια ιδιωτική εταιρεία η οποία θα δίνει τις πληροφορίες και θα εξασφαλίζει το ώστε να εφαρμόζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις από όλα τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη ε, και είναι θέμα εθνική αρμοδιότητα σε μεγάλο βαθμό και δεν μπορώ να το σχολιάσω περαιτέρω. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Παλάκη. <clears throat> E, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Υπουργέ, για αυτή την ενδελεχή λεπτομερέστατη απάντηση. Βλέπω ότι η Σουηδία πραγματικά ανησυχεί ιδιαίτερα και ενδιαφέρεται για την πνευματική διάσταση των αγωγών και το τι συμβαίνει στις χώρες της Βαλτικής. Να επαναλάβω όμως, τέτοιου είδους ζητήματα, τέτοιου είδους προβλήματα δεν πρέπει ποτέ να υποτιμώνται ως προς τις διαστάσεις τους. Ποτέ δεν θα είναι αρκετή η προσοχή που θα τους αποδίδουμε. Τόσο σημαντικά είναι. Ε, απευθύνω λοιπόν έκλεισε προς τη Σουηδία να παρακολουθεί στενά την κάθε εξέλιξη, το κάθε παραμικρό βήμα πρόοδου που μπορεί να επιφέρεται σε αυτό το, στην οικοδόμηση αυτού του αγωγού. Ευχαριστώ. Ε, θα σας καθησυχάσω. Μα το κάνει αυτό ήδη η Σουηδία παρακολουθούμε και γνωρίζουμε πόσο ευαίσθητο είναι το περιβάλλον ε, στην Βαλτική θάλασσα και γνωρίζουμε τους κινδύνους που συνεπάγονται διάφορα τέτοια προγράμματα και γι' αυτό έχουμε θέσει αυστηρότατες περιβαλλοντικές απαιτήσει γι' αυτό το πρόγραμμα ε, και εξετάζονται οι απαιτήσει από όλες τις συναρμόδιες αρχές. Ε, δεν, είναι, δεν μιλάμε μόνο για σουηδικό θέμα, δεν είναι δική μας επικράτη. Γι' αυτό σας μίλησα για τη σύμβαση ΕΣΠΟ του ΟΗΕ, ε, στην οποία βασιζόμαστε για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε. Ε, δεν κάνουμε πολιτική και οικονομική αξιολόγηση. Ε, το σουηδικό κράτος βασίζεται σε απαιτήσει που προβλέπονται σε αυτή τη σύμβαση. Σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Και τώρα επόμενη ερώτηση. Τώρα επόμενη ερώτηση, ερώτηση της κυρίας Τσίκαου για την κατάρριξη των φραγμών στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Ε, θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται στις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δικαίωμα λοιπόν των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μένουν και να εργάζονται σε ένα άλλο κράτος της Ένωσης. Ε, στις 9 Μαρτίου 2009 το Συμβούλιο απίθυνε πρόσκληση στα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν ε, τους κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ε, και ε, παρακολουθούμε την εφαρμογή ε, ως προς αυτούς τους φραγμούς. Ε, θα πρέπει να έρθουν οι φραγμοί στην τρίτη φάση εφαρμογής ε, εάν δεν διαπιστωθούν σοβαροί κίνδυνοι παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας εσωτερικής αγοράς. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εξετάσουν την κατάσταση και στη σχέση με τις τρίτες χώρες, γιατί θα πρέπει να καλυφθεί και η μεταβατική περίοδος ε, για όσους διέμεναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης θέματα οικογενειακής επανένωσης. Χρειαζόμαστε ευελιξία στους ε, κανόνες ε, φυσικά και τα κράτη-μέλη ε, λένε ότι θέλουν, τα νέα κράτη-μέλη θέλουν να αυξηθεί η πρόσβαση των πολιτών τους στις, αγορά, στις αγορές των υπολείπων κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Νοέμβριο του 2008 είχαμε και την ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της κατάστασης μετά τη διεύρυνση και διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι πολίτες από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, και των υπολείπων νέων κρατών μελών ε, είχαν πρόσβαση στις ε, αγορά εργασία στη χώρα ε, υποδοχή και ότι ενίσχυσαν την οικονομική ανάπτυξη σε αυτέ τι χώρε. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα και μετά την διεύρυνση δεν σημειώθηκε καμία παρεμπόδιση τη ομαλή λειτουργία τη εσωτερική αγορά και ούτε και πρόκειται. Υπάρχουν ε, κανόνες ε, για τον περιορισμό της πρόσβασης τους ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της αγοράς ε, και χρειάζεται κάποια προσαρμογή ορισμένες φορές στην αγορά εργασίας για μια μεταβατική περίοδο για να μην ενισχυθεί η παράλληλη οικονομία. Η κινητικότητα οδηγεί σε περισσότερες θέσεις απασχόλησης και σε καλύτερη αντίδραση των αγορών σε καταστάσεις οικονομικής κρίσης. Επίσης βοηθάει στην καταπολέμηση αποξένωσης και της ευτόχειας. Ε, τώρα για την μεταβατική περίοδο, αυτή για την οποία μας ε, ρωτάτε, φυσικά τα κράτη-μέλη μπορούν να διατηρήσουν τους περιορισμούς μέχρι να λήξει η τρίτη φάση της μεταβατικής περίοδου. Το Συμβούλιο θεωρεί βέβαια ότι η οικονομική κρίση που βιώνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως λόγος ε, για να συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυτοί οι μεταβατικοί κανόνες και Μπορεί να είναι δύσκολο οι ε, εργοδότες να αντιμετωπίσουν ναι, την ε, προσφορά εργασίας ακόμη και από τους πολίτες ε, της δικής τους χώρας. Ε, τον Ιούνιο του 2009 το Συμβούλιο ε, έλαβε υπόψη την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση και ενημερώθηκε από την Επιτροπή ότι ε, την 1η Μαΐου του 2009 τρεις από τις 10 χώρες είχαν κοινοποιήσει σοβαρούς κινδύνους για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Ε, και ε, ζητούν να διατηρηθεί η μεταβατική κατάσταση ενώ παραδείγματος χάρη το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να υπάρχει ε, καταχώρηση των εργαζομένων Ε, επιφυλασσόμεθα λοιπόν ε, και θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση κυρίως ε, στα κράτη-μέλη που συνεχίζουν να εφαρμόζουν αυτούς τους μεταβατικούς κανόνες. Ευχαριστούμε κυρία Τικά. Ευχαριστώ Υπουργέ. Να σας ρωτήσω αν στις προτεραιότητες της Προεδρίας, στο δικό σας χρονοδιάγραμμα, έχετε προβλέψει δράση για να προσπαθήσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη που διατηρούν φραγμούς και περιοριστικά μέτρα στην ελεύθερη ε, κυκλοφορία των εργαζομένων ε, να τα παροτρύνουμε να τα άρουν. Και μια δεύτερη ερώτηση. Η πρόταση για την άρξη των φραγμών. Δεν θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού, κατά τη Σουηδική Προεδρία. Υπουργέ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε. Ε, Ευχαριστώ. Κυρία Βουλευτά, η Γαλλική, ε, Τσεχική και Σουηδική Προεδρία στα συμπεράσματά τους δήλωσαν ότι ήταν πολύ ευρυγητική για την Ευρωπαϊκή Ένωση η διεύρυνση και σήμανε οικονομική ανάπτυξη. Δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι έχουν μεγάλες τρευλώσεις ε, οικονομικού τύπου. Έχουμε μηχανισμούς που σε τακτά χρονικά διαστήματα ε, ελέγχουν όλα αυτά τα στοιχεία και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε να ζητήσουμε κάθε φορά από τα κράτη-μέλη να ε, λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αρθούν οι διακρίσεις καθώς και η νομοθεσία που οδηγεί σε διακρίσεις για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό και τα εργατικά χέρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είστε ε, βέβαια ότι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχουμε τακτικά αυτά τα θέματα. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ρωτάει η ε, κυρία Τσικάου από τη Σκοπιά της ε, ε, από, ως μια χώρα που είναι προέλευσης αυτών των εργαζομένων. Ενώ στην Αυστρία έχουμε πρόβλημα εάν ανοίξουμε μέσω τα σύνορα για όλους τους εργαζομένους. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές εισοδήματος και ε, βλέπουμε να συρρυκνώνεται η αγορά εργασία. Αν αυξηθεί η μετανάστευση θα σημαίνει αυτό τεράστια επιβάρυνση τη αγορά και κοινωνικέ εντάσει που δεν τι επιθυμεί κανεί από εμά. Ερώτηση λοιπόν. Αυτά τα προβλήματα που τίθενται για την Αυστρία ή για τη Γερμανία τα καταλαβαίνετε, τα αναγνωρίζετε, τα γνωρίζετε, είστε πρόθυμοι και προβλέπετε ε, να προτείνετε συγκεκριμένες λύσεις. Ευχαριστώ. Η Υπουργός έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι όλα τα κράτη-μέλη πλήττονται από ανεργία και οικονομική κρίση. Μπορεί τα αριθμητικά στοιχεία να ε, διαφέρουν από χώρα σε χώρα, αλλά όλες οι χώρες έχουν πληγεί. Υπάρχουν μεταβατικές ε, ρυθμίσεις στην Αυστρία δικαιολογημένες και υπάρχει επίσης δυνατότητα παράτασης για συγκεκριμένα θέματα με αιτιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς την κατάσταση στην Αυστρία, οφείλω να το ομολογήσω. Μπορεί να έχετε περισσότερα προβλήματα από άλλα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της μας λέγει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να δείχνει ότι η ελευθερία ε, στη ε, κυκλοφορία διαταράσσεται ή στρεβλώνεται. Και η ίδια μου χώρα, η Σουηδία, που έχει πολύ ψηλή ανεργία, δεν έχει διαπιστώσει να υπάρχει σχέση ανάμεσα στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την αύξηση της ανεργίας. Έχουν απορροφηθεί χωρίς προβλήματα. Περνάμε, ευχαριστώ, στην επόμενη ερώτηση τώρα του κυρίου Χουντή. Παρενόχληση της Τουρκίας σε βάρος εναέριων μέσων της Υπηρεσίας Ελέγχου Εξωτερικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Frontex. Παρακαλώ. Eh, Πρόεδρε, το Συμβούλιο έχει επίγνωση αυτών των γεγονότων που αναφέρει ο αξιότιμος βουλευτής. Η Προεδρία θέλει να πει ότι η Τουρκία ως υποψήφια χώρα πρέπει να σέβεται τις αξίες και τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στις συνθήκες. Πρέπει να υπάρχει καλή γειτονία και ειρηνική επίλυση των διαφορών. Αυτό ε, ε, είναι μια απέτηση καταλητική σημασία για όλες τις υποψήφιες χώρες στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και σας παραπέμπω και στα αντίστοιχα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Έχουμε παρακαλέσει την ε, ε, Τουρκία να μην ε, δημιουργεί προστριβές και να επιδιώκει τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Το θέμα των σχέσεων καλής γειτονίας συστηματικά αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 19 Μαΐου στο Συμβούλιο με την Τουρκία και στη συνάντηση της Τρόικα τον Ιούλιο με τους πολιτικούς διευθυντές της Τουρκίας αναφέρθηκε το ζήτημα. Γι' αυτό το συγκεκριμένο αεροπλάνο του Frontex Ήθελα να σας πω ότι συντονίζει πολλές κοινέ επιχειρήσεις ε, ο Frontex ε, και είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό το θέμα για τα θαλάσσια και τα ενέργεια σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε και τον Ποσειδώνα. Αμφιτρίωνας είναι η Ελλάδα σε αυτό το πρόγραμμα. Μιλάμε για ανθρώπους που έρχονται από την Βόρεια Αφρική και προσπαθούν να πάνε στις ακτές της Ελλάδας. Φυσικά γνωρίζετε την κατάσταση. Επίσης μιλάμε για πώς απόσπασης ε, ε, αξιωματικών συνδέσμων που θα τοποθετηθούν σε νησιά, παραδείγματο χάρη τη Ελλάδα, για την συνεργασία ανάμεσα στο Frontex και τι αρμόδιε τουρκικέ αρχέ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει για τη μέθοδο εργασία. Αυτό είναι θετικό. Ε, και μια ενδεχόμενη συμφωνία θα καλύπτει και την ανταλλαγή πληροφοριών και τη δυνατότητα των τουρκικών αρχών να συμμετάσχουν στι κοινέ επιχειρήσει του Frontex. Αυτό είναι σημαντικό για την καταπολέμηση τη λαθρομετανάστευση ε, και την βελτίωση των σχέσεων καλή γειτονία. Σα ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Χουντή. Πρόεδρε, <clears throat> κυρία Υπουργέ, αφού σα επαναλάβω για άλλη μια φορά την εκτίμησή μου για τη φιλότιμη προσπάθεια που κάνετε για να δίνετε απαντήσει σε αυτά που ρωτάμε, επιτρέψτε μου να σα πω ότι από αυτά που μου είπατε, μου λέτε το περιστατικό σα είναι γνωστό, με την Τουρκία συνεργαζόμαστε, αλλά δεν είναι σαφή απάντηση και γι' αυτό εστιάζω και επαναλαμβάνω την ερώτηση αν πράγματι κατά την αποστολή Frontex έγιναν παραβιάσεις του εναέριου χώρου της τουρκίας όπως η ίδια ισχυρίζεται. γιατί το λέω αυτό; διότι μέσω από αυτές τις διαδικασίες διερευνάται αν η τουρκία αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της ελλάδας. συμπληρωματικά σας λέω ότι ο αναπληρωτής εκτελεστικός διευθυντής της frontex ο κύριος φερνάντες σε πρόσφατη επίσκεψη στην ελλάδα ισχυρίστηκε ότι δεν γίνονται τέτοιες παραβιάσεις παραπέμποντας το θέμα σε αναφορές των πιλότων. επανέρχομαι λοιπόν υπάρχουν ή όχι οι παραβιάσεις τις οποίες ισχυρίζεται η τουρκία με βάση την αποστολή frontex και τι κάνετε απέναντι σε αυτό. Πρόεδρε, είναι ε, πολύ δύσκολο για τη Σουηδική Προεδρία να ε, αποφασίζει πότε ε, υπάρχει παραβίαση και πότε όχι. Έχουμε γνωρίζουμε την ανησυχία πολλών Ελλήνων συναδέλφων και έχουμε ε, ε, προάγει τον διάλογο με τις τουρκικές αρχές για αυτό το ζήτημα και ενθαρρύνουμε πάντοτε σε όλες τις επαφές ε, τις τουρκικές αρχές να διατηρούν αυτές τις σχέσεις καλής γειτονίας αλλά για μια προεδρία είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρίνει αν συνιστά κάτι η παραβίαση ή όχι γιατί είναι θέμα διεθνούς δικαίου και θέμα διμερών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Κυρία Μόρβάη, συμπληρωματική ερώτηση. Γι' αυτό το θέμα όμω έχετε ζητήσει το λόγο. 30 δεύτερα έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, διαβάζετε τη σκέψη μου. Έτοιμη μου να, να ζητήσω το λόγο για να ζητήσω συγγνώμη που θα πάρω άλλα 20 δευτερόλεπτα από το χρόνο σας από την τόσο ζωντανή πολυπληθή δημοκρατική συζήτηση για ένα τέτοιο άσχετο θέμα όπως είναι η πολιτική κρατούμενη και η αστυνομική βία σε ένα κράτος βέλος. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όταν έχετε συμπληρωματική ερώτηση, μπορείτε άλλη ερώτηση να την υποβάλλετε γραπτός με την κανονική οδό και να απαντηθεί, ε, αν χρειαστεί να απαντηθεί. Υπάρχουν πολλά μέλη που θέλουν να δουν τις ερωτήσεις του σήμερα να απαντώνται και παρακαλώ λίγο σεβασμό για να έχουμε τακτική διαδικασία εδώ. Λοιπόν, Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Είναι παρόν ο συντάκτης. Απουσιάζει ο κύριος Βανέκε. Η ερώτηση της κυρίας Μαγκίνες είναι η επόμενη. Λοιπόν, αναθεώρηση του κανονισμού υπαριθμών 1 κάθετος 2005. Κύριε Υπουργέ, και υποθέτω, υποπτεύομαι ότι είναι η τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ και ευχαριστώ την κυρία Μαγκίνεσε για την ερώτηση. Φυσικά και εμείς ανησυχούμε για την ευημερία των ζώων όπως η αξιότιμη βουλευτή. Έχουμε ήδη απαντήσει μια παραπεριφερή ερώτηση της κυρίας εκείνη το Σεπτέμβριο και ε, ο στόχος της Προεδρίας είναι να προάγει τον διάλογο για την ευημερία των ζώων. Συνιστά προτεραιότητα αυτό για την Προεδρία μας. Ε, στις 7 Σεπτεμβρίου ενημερώθηκε από την Επιτροπή το Συμβούλιο σχετικά με ένα σχέδιο πρότασης ε, ε, την αναθεώρηση του κανονισμού 1-2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά και αναμένεται σε λίγο καιρό ε, και συμφωνούμε ότι χρειάζονται νέα μέσα για καλύτερο έλεγχο, καλύτερη επιθεώρηση των διεθνών μεταφορών ζώων των ζώων. Παραδείγματο χάρη ένα σύστημα παρακολούθηση με δορυφόρο. Ένα τέτοιο σύστημα θα διευκόλυνε την εποπτεία από πλευρά των αρχών των κρατών μελών, γιατί πολύ δύσκολα μπορεί κάποιο να καταδείξει ε, ότι υπάρχουν ατέλειε, παραδείγματο χάρη, με τα μέσα που χρησιμοποιούμε σήμερα. Ε, και η αναθεώρηση αυτού του κανονισμού σημαίνει ότι θα υπάρχει καλύτερη προστασία των ζώων ε, διότι θα προβλέπετε ποια είναι τα εμπλεκόμενα μέρη και αναγνωρίζετε ποια είναι η ευθύνη του καθενός. Ενισχύουμε τα μέτρα ε, για τις ε, επιθεωρήσεις και υπάρχουν αυστηρότεροι κανόνες ε, για την μεταφορά. Κάποιες επιτυχίες δεν καλύπτονται όμως από τον κανονισμό. Παραδείγματο χάρη ανώτατος αριθμός ταξιδιών και απαιτήσει για τα ζώα. Βάσει του άρθρου 32 του κανονισμού θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή έκθεση ε, ρύθμιση που θα αρχίσει να ισχύει μετά από τέσσερα χρόνια και μόλις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει την πρότασή της ε, θα ε, ακολουθήσει η επεξεργασία του θέματος από το Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πάντως ε, για το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται για το, ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ για την εκτενέστατη απάντηση. ανησυχώ κι εγώ για την ευημερία των ζώων, αλλά θέλω ένα κανονισμό ρεαλιστικό που αφορά το εμπόριο στα ζώα, ε, που να είναι θέμητο και με το σωστό έλεγχο. Δεν χρειαζόμαστε επιπλέον ρυθμίσει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σωστή εφαρμογή τη κείμενη νομοθεσία. και ε, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σα, ε, για την αυσίπλοη και τα λοιπά. Α, δύο λόγια μόνο για τη μεταφορά ύπων. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει πρόβλημα, δεν εφαρμόζονται σωστά οι κανονισμοί. Δεν ξέρω ίσως να θέλετε να το σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Thank you, Madam Chair. I am not... Ευχαριστώ. Όχι, δεν είμαι ε, αρμόδια και εμπειρογνώμων στα υποειδή. Ε, σας ευχαριστώ για αυτά που λέτε, το σημειώνω. Είναι αρκετά συχνό αυτό το φαινόμενο να χωλαίνει η εφαρμογή. Δεν χρειάζεται πάντα νέους κανονισμούς κάτι, η νέα ρύθμιση. Όταν έρχεται μια πρόταση, εμείς τη μελετούμε, την αξιολογούμε και βλέπουμε αν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον μέτρα ή όπως είπατε και εσείς και υπενήσεστε, ε, μόνο ενίσχυση της εφαρμογής και τήρησης των κανόνων και των νόμων. Θα επανέλθουμε μόλις έχουμε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Κέλλη έχει συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε η κυρία Μαγκίνες, συνάδελφός μου. Ξέρετε ότι η Ιρλανδία εξαρτάται πάρα πολύ από την υπερπόντια μεταφορά ζώων και ε, είναι απαγορευτικό το κόστος πολλές φορές για τον κλάδο. Όταν κάνετε την αθεώρηση αυτά θα τα λάβετε υπόψη, γιατί αν δεν έχουμε μεταφορά ζώων των ζώων, τότε μπορεί να κλείσουν πολλά εργοστάσια και πολλοί κόσμος να μείνει στην ψάθα. Ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίες για την Ιρλανδία αφού είναι και νησί και πόσο εξαρτάται. Ε, αλλά εδώ βεβαίω ανησυχούμε βαθύτατα και υπάρχει και πίεση των πολιτών να σκεφτούμε και την ευημερία των ζώων. Να δούμε λοιπόν, να αξιολογήσουμε τι έχει γίνει, ε, αν τα πράγματα εφαρμόζονται σωστά, αν χρειάζεται επιπλέον νομοθεσία, ή μήπω ε, να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη πριν προχωρήσουμε σε νέα νομοθεσία. Θα συζητούμε με τα κράτη-μέλη και όλα τα κράτη θα έχουν την ευκαιρία να ε, διαβιβάσουν ε, τις απόψεις τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Είχατε την καλοσύνη να πείτε ότι θα δεχτείτε δύο ακόμα ερωτήσεις γιατί είχαμε δύο μέλη παρόντα. Ο κύριος Τούσας και ο κύριος Κέλλη θα απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Ο κύριος Τούσας ρώτησε για την άσκηση ηλεκτρονικού φακελώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αποχωρήσει ο κύριος Τούσας. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ε, κρίμα. Ο κύριος Σκέλη τότε για ένα χαρτοφυλάκιο ε, αθλητισμού. Και θα είναι η τελευταία ερώτηση. Χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον Αθλητισμό. Παρακαλώ. Εδώ είστε, ναι. Ναι, ήταν ο δεύτερο φακελό μου, πρέπει να το κοιτάξω. Κοιτάξτε, ο αθλητισμό είναι ένα θέμα που μα απασχολεί στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο σήμερα. Και όπω σωστά εντοπίζει ο κ. Κέλλη, όταν τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα, θα προβλέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομική βάση που θα επιτρέπει να συνεισφέρουμε στην προώθηση του αθλητισμού στην Ευρώπη και τα σχετικά ζητήματα, λαμβάνοντα υπόψη την ιδιαίτερη φύση του αθλητισμού, τι υποδομέ του, ε, τι ε, θεωρητικέ δραστηριότητε και την κοινωνική του λειτουργία και συμβολή. Ωστόσο, το Συμβούλιο δεν μπορεί να τοποθετηθεί για την εσωτερική διοργάνωση της ε, Επιτροπής, της Μελλοντικής Επιτροπής. Το τι θα γίνει με τη συνθήκη θα είναι θέμα του Προέδρου της Επιτροπής. Νομίζω ότι ο αθλητισμός και η υγεία πηγαίνουν χέρι με χέρι. Οι αθλητικές δραστηριότητες επίσης προωθούν την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία, την προσωπική ανάπτυξη, την, την ορίμανση και είναι και ψυχαγωγία. Γιατί και στους ποδοσφαιρικούς ομίλους και στα διεθνή πρωταθλήματα βλέπουμε πως ε, το πνεύμα του αθλήστε επηρεάζει θετικά. Το ίδιο και η κοινωνική υγεία, η διαφύλαξη των δημοκρατικών αρχών. Η Σουηδική Προεδρία θεωρεί ότι η πολιτική του αθλητισμού είναι καταρχά όμω εθνικό ζήτημα. Πρέπει να είμαστε λοιπόν προσεκτικοί με νέε προτάσει και προγράμματα τα οποία θα πολλαπλασιαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μπορεί να βλάψουν ήδη εύρωστα προγράμματα τα οποία η κοινωνία των πολιτών έχει θέσει εφαρμογή εδώ και χρόνια. Σα ευχαριστούμε, κύριο Σκέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την απάντηση στην ερώτησή μου. Ήσασταν ιδιαίτερα διεξοδικοί. Μιλήσατε πολύ σωστά για τι αξίε του αθλητισμού, ιδίω την διάσταση τη υγεία. Είμαι βέβαιο ότι όταν, θέση, όταν έχουμε την συνθήκη τη Λισαβόνα θα φροντίσουμε ο αθλητισμό να έχει τη θέση που αξίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάλληλη προβολή. Κυρία Μαγκίνε, θέλετε τον τελευταίο λόγο. Μια ερώτηση, γιατί ο κύριο Κέλλη είναι πολύ ντροπαλό δεν είπε ότι ήταν πρώην πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου των Γελικών και προωθούσε την, ε, τον αθλητισμό στην Ιρλανδία. Γι' αυτό ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τα σπορ και τον αθλητισμό. Ήθελα να το ξέρετε. Σας ευχαριστούμε που μας το επισημάνατε. Με αυτή την ευχάριστη παρατήρηση κλείνουμε τη συζήτηση. Οι ερωτήσει που δεν προλάβαμε να δούμε σήμερα θα απαντηθούν γραπτώ. Σα ευχαριστούμε, Υπουργέ. Δύο ενημερωτικά στοιχεία. Η συνάντηση στις 5 στις 5 Οκτωβρίου των νομικών υποθέσεων, της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων αποφάσισε ότι είναι απαράδεκτο η κοινοβουλευτική ασυλία του κυρίου Φιόρε να έρθει.